επιτροπές έχουν εκινήσει τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 69C, παράγραφος 1 του κανονισμού. Στη ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Δυνάμει του άρθρου 69C, παράγραφος 2 μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι αύριο της, την 4η Ιουλίου στις 12 το βράδυ να εκκινηθεί η διαδικασία διαπραγματεύσεων. Εάν δεν υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, στην προγενέστερη προθεσμία οι επιτροπές μπορούν να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις.